Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ζήτησε μία ερμηνεία του άρθρου, ενός άρθρου του κανονισμού 1896-2006. Η ερμηνεία αυτή θα εγκριθεί αν μέσα σε 24 ώρες καμία πολιτική ομάδα ή αριθμός βουλευτών, όπως ορίζεται από τον κανονισμό, δεν θα